rapporteur is ready and... Do we have a thing to make clear that we're starting somewhere? Yeah, you have a gavel. Oh, that's now. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I uh, suggest we starting. Καλό σας απόγευμα. Να θα αρχίσουμε παρόλο που δεν είναι εδώ όλα τα μέλη. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη διότι ο κύριος Σαφάρνο του οποίου η πτήση Ακυρώθηκε, δεν θα μπορέσει να έρθει. Και έτσι θα μοιραστούμε την προεδρία, θα μοιραστώ εγώ την προεδρία με τον κύριο Ταβάριτς. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Σχόλια παρακαλώ. Όχι. Δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών 18-19 Φεβρουαρίου. Που υπάρχουν και στα αγγλικά. Σχόλια, όχι. Ωραία. Μερικές ανακοινώσεις. Υποσχέθηκα στον κύριο Σμιτ να μπορεί να μιλήσει, να προσιάσει κάτι από αυτού του σημείου, επειδή θέλει, πρέπει να φύγει νωρίτερα. Μήπως κύριε Σμιτ θέλετε τώρα να μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημα μου έχει σχέση με τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 18 Φεβρουαρίου. Στο σημείο 3 λέει επιλογή των υψηλόβαθμων στελεχών οι οποίοι θα υποβάλουν συστάσεις στην Επιτροπή ΚΡΙΜ. Στην Επιτροπή μας. Ε, ξαφνιάστηκα όταν είδα ότι οι σοφοί συντονιστές μας αποφάσισαν να επιλέξουν μόνο <laughs> πέντε άντρε. και μάλιστα τόσο κοντά στην ε, ημέρα ε, που γιορτάζουμε τις γυναίκες. Ε, πέντε άντρε λοιπόν επιλέχθηκαν ως υψηλόβαθμα στελέχη. Πολύ παράξενο αυτό. Κάποιος μπορούσε να πει ότι δεν υπήρχαν επιλέξιμες κυρίες, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, διότι είχα εγώ ο ίδιος προτείνει μία κυρία. Τώρα, εάν θέλουμε την ε, ισότητα των φίλων ή τη διάσταση τέλο πάντων του φίλου να τη σεβαστούμε, ελπίζω να μπορεί να αλλάξει αυτό το στοιχείο. Είναι ένα αρνητικό μήνυμα από την Επιτροπή μας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, εμείς φταίμε είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Όλες οι πολιτικές ομάδες και η δικιά μου έχουν υποβάλει ε, ονόματα που είναι όλα ανδρικά, είναι όλο άρενες. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες επιλέξιμες εκτός από τους άνδρες συναδέλφους. Και ε, το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα το βράδυ που συνεδριάζουν οι συντονιστές και αυτοί είναι που αποφάσισαν εν πρώτης, θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ο κύριος Σμιτ, για να είμαστε σαφείς. Εγώ έχω να προτείνω μία κυρία, ένα γυναικείο όνομα. Α, τότε λέει ο πρόεδρος, δεν με είχαν ενημερώσει σωστά. Θα το συζητήσουμε λοιπόν το βράδυ και αν συμφωνείτε όλοι θα μπει ε, στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών σήμερα το βράδυ για προς αναθεώρηση ή δυνατόν. Εν συνεχεία, όπως ε, ίσως ξέρετε, είμαστε στο διαδίκτυο, ζωντανά αυτή η συνεδρίαση και τις 5.30 και κλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσουν οι συντονιστές και θα, θα πάρουν αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων. Αυτά λοιπόν επί του σημείου 3. Τώρα θα προχωρήσουμε στο σημείο 4, εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Και χρειάζομαι απαρτία. Δεν νομίζω ότι έχουμε απαρτία αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Προτείνω να αρχίσουμε τη συζήτηση και να περιμένουμε μέχρι ότου έχουμε απαρτία. Τρία μέλη χρειαζόμαστε ακόμα για απαρτία. Αν μπορείτε να ειδοποιήσετε κάποιον συνάδελφο να έρθει, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάρουμε την απόφαση τώρα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, μία παράκληση. Επειδή εμείς έχουμε υποψήφιο, προτείνουμε υποψήφιο, τον Αντιπρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Λιάννα Λιώτοβα που κάθεται πίσω μου θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν μπορέσετε να καλέσετε τρία μέλη ακόμα να έχουμε την απαρτία, διότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία της εκλογής αντιπροέδρου, του πρώτου αντιπροέδρου. Θα ήθελα λοιπόν ή δυνατόν ε, να καλέσουμε τρία μέλη πριν φύγει κάποιος για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκλογή. Ο πρόεδρος, ναι, οι υποψηφιότητες είναι σαφείς, έχουν υποβληθεί από τις πολιτικές ομάδες. Ίσως η κυρία υποψήφια θέλει να μας ε, έχει κάτι να πει, αν συμφωνείτε με αυτήν την υποψηφιότητα, <laughs> νομίζω είναι η μόνη. Δέχεστε, δέχεστε την υποψηφιότητα σας. Ευχαριστώ για τον διορισμό. Συμφωνώ και περιμένω την ψήφο των συναδέλφων σας. Well, Ωραία, έχουμε κάνει λοιπόν τα πρώτα δύο βήματα και τώρα θα κάνουμε την, ε, θα ψηφίσουμε όταν μπορέσουμε να έχουμε απαρτία κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Φτάνουμε τώρα στο κύριο θέμα της σημερινής διάταξης που είναι η παρουσίαση και συζήτηση της ε, προσωρινής, ε, του προσωρινού σχεδίου ε, γνωμοδότησης του σχεδίου έκθεσης και θα ζητήσω τον κύριο Γιακολίνο που είναι εισηγητής να μας μιλήσει το πολύ για 20 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρκεστώ το, στο χρόνο που μου ορίζεται. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δραστηριότητα που προσπαθώ να σκιαγραφίσω συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πολιτικές ομάδες, τους σκιώδεις, τους συντονιστές και τη γραμματεία για αυτή τη δραστηριότητα την οποία προωθήσαμε και προωθούμε με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη ένταση δραστηριοτήτων με βάση την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποβάλαμε τρία έγγραφα για το οργανωμένο έγκλημα, για τη διαφθορά και για την ανακύκλωση χρήματος. Επίσης, ορίσαμε τον γενικότερο μας στόχο, δηλαδή να προσεγγίσουν, να υπάρχει καλύτερη προσέγγιση της εσωτερικής ένομης τάξης των κρατών μελών, έτσι ώστε να υπάρχει μία ομογενοποίηση ε, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν ε, ορισμένα αριθμητικά στοιχεία για τη μέτρηση ενός ε, φαινομένου που δεν είναι μόνο κοινωνιολογικό, αλλά ενέχει και εγκληματικά στοιχεία στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Οι πρόσοδοι αυτοί φτάνουν στο 3,6% του ΑΕΠ. 388 δις δολάρια αποτελούν το ύψος του, των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου, ενώ 320 δις προέρχονται από τα ναρκωτικά και από ανακυκλωμένο χρήμα. Μιλάμε για ένα 2 έως 5% του παγκοσμίου ΟΑΕΠ. Μιλάμε για 650 δις 550 ε, εκατομμύρια. Έτσι βλέπουμε τον αριθμό των στοιχείων που αφορούν τα εγκληματικά στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας. Στην Ευρώπη υπάρχουν 3.600 οργανωμένες ε, ομάδες εγκλήματος και μιλάμε για 120 δις δολάρια. Αυτό είναι το, ε, αυτός είναι ο τζίρος και 12 δις είναι το συνολικό κόστος από τη διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για τα πιο προσοδοφόρα στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματος. Τα 11 δις, 11 δις σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση σιγαρέτων και 1 δις, 1 δις εκατό αποτελεί τον τζίρο των ε, παραχαραγμένων προϊόντων. 100 δις ετησίως είναι ο υπολογισμός για την φοροαποφυγή και 1,5 δις αφορά απάτες από παράνομη χρήση πιστοτικών καρτών. Πρόκειται λοιπόν για πολύ σημαντικά στοιχεία που έχουν ε, μεγάλη επίπτωση στον οικονομικό ιστό. Στόχος αυτής της έκθεσης και αυτής και της ενδιάμεσης που ορίσαμε με τη συνδρομή των άλλων πολιτικών ομάδων έγκυται στο να υπερασπιστούμε τους έντιμους πολίτες να πιστεύουν στο δημοκρατικό σύστημα και να προωθήσουμε τους έντιμους επιχειρηματίες και τη σχετική οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία νομοθετική προσέγγιση που θα συμπληρώσουμε μέχρι το τέλος του έτους με την έγκριση του εγγράφου αυτού. Επίσης, η ε, δουλεμπορία αντιμετωπίζεται διεθνώς. Μας ενδιαφέρει και η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η παράνομη διακίνηση τσιγάρων. Βλέπουμε μια διαχρονική αύξηση αυτής της εγκληματικότητας για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφορά και το ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματος θα πρέπει να υπάρχει, να προβάλλουμε ένα σύστημα κατάσχεσης, οι μαφιόζικες οργανώσεις να μην μπορούν να συμμετάχουν σε ανάθεση δημοσίων έργων, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και συνεργασία για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβέρνοχώρο και στα παράκτια. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί. Οι εγκληματικές οργανώσεις κινούνται εκεί που υπάρχουν μεγάλοι πόροι, επιχειρήσεις, κατανομή πλούτου και ιδιαίτερα ως προς τα παραχαραγμένα είδη εκίδρα το οργανωμένο έγκλημα και εκπροσωπεί όχι όλα τα κράτη-μέλη, αλλά όλα τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία στον δικαστικό τομέα, στον αστυνομικό τομέα, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε μια πιο υπεύθυνη πολιτική και μια πολιτική που να αναλάβει τις ευθύνες της ολοκληρωτικά. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες κυρώσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα, καθώς και μία άλλη αντιμετώπιση του θέματος από τη δημόσια διοίκηση. Υπάρχει έντονη γραφειοκρατία πολλά χαρτιά που περνάνε από το ένα γραφείο στο άλλο και πολλοί φορείς πρόληψης με υπέρογγη γραφειοκρατία, κάτι το οποίο δεν βοηθά ιδιαίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιτάξουμε κάτι άλλο. Να υπάρχει ένα σύστημα αυστηρών κυρώσεων με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και ένας σύστημα το οποίο να μην ε, παραγράφει το έγκλημα. Να υπάρχει εποπτεία και εγγύηση των δικαιωμάτων του υποδίκου, αλλά παράλληλα δεν θα πρέπει να, υπάρχει, να οδηγούμεθα σε ατιμορρησία με βάση μακροχρόνιες ε, διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου. Ε, επίσης, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εποπτεία. Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερα white lists, δηλαδή επιχειρήσεις, ε, καταλόγους μάλλον με σύνομες εταιρείες ή επιχειρήσεις. Και εδώ μιλώ για, την, για ένα σύστημα ανακύκλωσης της διακυβέρνησης των ε, τραπεζών. Και αυτό αφορά και τα εμπορικά επιμελητήρια, τα οποία μπορούν να αναλάβουν ευθύνη, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει υποψία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το οποίο έχει διεθνικό χαρακτήρα. Όσο αφορά την απάτη, απάτη ταυτότητας, απάτη έναντι των φορολογικών αρχών ή των ευρωπαϊκών αρχών, ίσως χρειάζεται μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, η οποία να διασφαλίζει τα σύνομα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτική αρχή, έτσι ώστε να μην υπάρχει match fixing και χρειάζεται διαφάνεια και σαφήνεια στις συναλλαγές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις τεχνολογίες εχμής για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, όπως είναι και το σχετικό σύστημα της Europol, καθώς και δορυφορικά συστήματα. Επίσης, ε, όταν υπάρχουν απατηλά στοιχεία στους υπολογισμούς, φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται. Εμείς θέλουμε δίκαιες φορολογικές αρχές που να λαμβάνουν υπόψη ότι αυτός που παράγει θα πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο αυτού που έχει παράγει. Επίσης, ε, οποιαδήποτε δραστηριότητα της ε, μαφίας ε, θα πρέπει να διώκεται σε όλα τα κράτη-μέλη διαφορετικά. Η ίδια και απόφαση του δικαστηρίου δεν θα την χάνει της ίδιας αντιμετώπισης. όπως ε, μπορεί να συμβεί ε, σε περίπτωση εφαρμογής σε άλλο κράτος από το κράτος προέλευσης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ε, μέτρησης των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το κάθε κράτος έχει φέρει υψηλή ευθύνη, μεγάλη ευθύνη. Οι δραστηριότητες της μαφίας υπάρχουν στα περισσότερα κράτη-μέλη, γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία με την Όλαφ και την Eurojust καθώς και την Europol. Χρειάζονται προγράμματα και τύπου έρασμους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και δημόσια διαφθορά καθώς και την διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, οι βουλευτές, εάν υποπέσουν σε κάποιο παράπτωμα, θα πρέπει να δεχτούν τις αντίστοιχες κυρώσεις και για πέντε χρόνια να μην έχουν την ε, πιθανότητα, την δυνατότητα μάλλον του εκλέγην και εκλέγεστε ιδιαίτερα σε περίπτωση διαφθοράς οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών παραπτωμάτων που άπτονται της δημόσιας διοίκησης. Προτείνουμε μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων επίσης και κυρώσεις αν υπάρχουν καταχρήσεις και κατασπατάληση. Στο θέμα της διαφθοράς θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση, να υπάρχουν εγγυήσει που να συνάδουν και να συμβαδίζουν με τους καιρούς που διανύουμε ως προσήτηματα διαφοράς, διαφθοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να πλήξουμε το έγκλημα γενικότερα και να πλήξουμε και παράνομες δραστηριότητες. δραστηριότητες. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να υπερασπιστούμε τα θύματα της μαφίας. Η υπεράσπιση επίσης των μαρτύρων. Αυτό προβλέπεται και στο τελικό μας κείμενο, αλλά θα δεχτούμε και τις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Επίσης θα πρέπει να πατάξουμε τους φορολογικούς παραδείσους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάπτοντας εμπορικές συμφωνίες, δεν πρέπει να ξεχνά ότι στην Ασία, στη Σιγκαπούρη, αλλά και αλλού ε, υπάρχουν φορολογική παράδεισοι και μια διαφορετική πραγματικότητα, όπου υπάρχει ένα match fixing. Τέλος, θα πρέπει να μην υπάρχει τέτοιος φορολογικός φόρτος των ΜΜΕ. Στην Ιταλία ανέρχεται στο 45% του κύκλου εργασιών. Θα πρέπει όμως να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν φορολογική παράδοση και στην Ευρώπη, όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να υπάρχει θέληση για ένα πρόγραμμα δράσης για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, την Κομισιόν, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ε, ανακύκλωσης βρώμικου χρήματος. Πολύ συχνά δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι σε τραπεζικά ιδρύματα. Γι' αυτό χρειάζονται επαρκείς κυρώσεις μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης των παράνομων δραστηριοτήτων όπως παράνομη διακίνηση τσιγάρων ή λαθρεμπορία. Λαθρεμπορία προσώπων. Με την συνδρομή λοιπόν των πολιτικών ομάδων τα καταφέραμε. Θα ήθελα ε, να, ευχαριστήσω τους άλλους δέκα από κοινού συντάκτες για την ενδιάμεση αυτή έκθεση την οποία έχω αναλάβει. Προσπαθήσαμε να συμπυκνώσουμε τη δραστηριότητά μας. θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγκάρσια προσέγγιση αντιμετώπισης των εγκληματικών οργανώσεων, των μαφιών και του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Την προηγούμενη εβδομάδα, Πρόεδρε, συναντήθηκα με τους Σκιώδης και μιλήσαμε για ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα μας κατευθύνει για να φτάσουμε σε ένα αίσιο πέρας. Έχουμε ορίσει και μία προθεσμία υποβολής τροπολογιών 25-26 Μαρτίου για να υποβληθούν οι τροπολογίες και λάβαμε υπόψη να εγκριθούν στις 18 Απριλίου στο Στρασβούργο για να γίνει ψηφοφορία στην ΚΡΙΜ την 3η ε, 23 Απριλίου και ψήφιση στην Ολομέλεια το Μάιο ή τον Ιούνιο. Πρόκειται για χρονικά διαστήματα που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την συμβολή των πολιτικών ομάδων. Συμφωνήσαμε με τους σκιώδεις να προτείνουμε τροπολογίες και μέσω κειμένων τα οποία να συμμερίζονται περισσότεροι του ενός. Τα πρώτα έγγραφα πριν από το ενδιάμεσο αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης από την Κομισιόν και είμαι πεπισμένος ότι αυτός ο καλός διαρθρωμένος διάλογος θα μας βοηθήσει μέσα στα πλαίσια αυτού του χρονισμού και η γραμματεία θα μπορέσει να μας βοηθήσει και να βοηθήσει τα 500 εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ στην υπόθεση και θέλουν μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη θέληση και αντιμετώπιση των εγκληματικών συστημάτων καθώς και των συστημάτων της μαφίας με μια μεγάλη θέληση, με μεγάλη θέληση. Περιμένω την αντίδραση των συναδέλφων και όπως σας είπα μπορούν να γίνουν διορθώσεις και συμπληρώσεις. Για να δούμε κατά πόσο η Επιτροπή μπορεί να συντάξει αυτό το πρώτο ιστορικό έγγραφο αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλήματος. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκφράζει τα 500 εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν εκ του σύνεγγι στο θέμα και θέλουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη αντιμετώπιση των εγκληματικών συστημάτων, της μαφίας και της ανακύκλωσης. Είμαι στη διάθεσή σας ε, για περαιτέρω διευκρινήσεις και ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την εντολή που λάβαμε εδώ και ένα χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιακολίνο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Όχι μόνο καλύψατε όλο αυτό το εύρο ζητημάτων που έπρεπε να καλύψετε, αλλά το κάνατε και μέσα στα 20 λεπτά που σα είχαμε αναθέσει. Είναι καλό λοιπόν να περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων. Τρει έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Ματιέ από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε χαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα των εργασιών του και την πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων που είχαμε κάνει στο παρελθόν. Πολύ ποιοτικό το έργο του λοιπόν και πρέπει να το συγχαρούμε. Δεν ισχύει πάντα εδώ στο Κοινοβούλιο αυτό. Μας παρουσιάζει λοιπόν ένα ιδιαίτερα πλήρες και περιστατωμένο σχέδιο έκθεσης, όπως είπατε και εσεί Πρόεδρε, με μια πολύ ε, ε, δεκπεριωτική ή μάλλον ε, πληρέστατη περιγραφή της κατάστασης με όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε τη μαφία, τη διαφθορά, την, το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Είναι αυτό το ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Επίσης, στο σχέδιο έκθεσης ε, βλέπουμε ότι με το άρθρο 183 της Συνθήκης της Λισαβόνας η Επιτροπή μπορεί να κάνει κάποιες προτάσεις ε, για να αναρμονίσει το ποινικό δίκαιο ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό γιατί, όπως είπατε, οι μαφίες υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και αν στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε κάποια μέλη δεν έχουν ε, επίγνωση της δράσης της μαφίας. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τη μαφία και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ της μαφίας της Ευρωπαϊκής και των μαφιών σε τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα είναι πραγματική μάστιγα, ιδίω ε, κατόπιν της ε, κρίση που βιώνουμε σήμερα. Είναι κάτι που υπογραμμίζετε κι εσείς στην έκθεσή σας. Ιδίω λοιπόν ε, σε συνθήκες κρίσης αναπτύσσεται γιατί βασίζεται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, ό,τι βρίσκεται στι δυνατότητε μα για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Α περάσω τώρα στο ξέπλυμα χρήματο. Αναφερθήκατε εκτενέστατα και σε αυτό. Αλλά και ε, σε ό,τι αφορά το εμπόριο ανθρώπων που είναι ένα ιδιαίτερα ε, βάναυσο έγκλημα. Έχετε δώσει κάποιες ε, πιθανές λύσεις σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της κατάρτισης ε, των αστυνομικών αρχών αλλά και των δικαστικών αρχών. Αναφερθήκατε σε έναν καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών οργανισμών, μίλησατε για την Eurojust, για την Europol, για την κατάρτιση μαζί με την SEPOL. Εξαιρετικά σημαντικό, αλλά και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Εισαγγελική Αρχή. Πολύ θετικά όλα αυτά. Θα μείνω εδώ. Να πω μόνο ότι προφανώς και θα στηρίξουμε την ε, έκθεσή σας που είναι ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη. Ε, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τους ε, σκιώδεις. Και εμείς σημειώσαμε και την ημερομηνία υποβολής καταθέσεων, αλλά δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε όπως και να έχει. Από την άλλη, μιλήσατε για τις 18 Απριλίου για την συζήτηση των εξέταση των τροπολογιών. Ίσως αυτό να συζητηθεί στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών, γιατί έχουμε εκείνο το πρωινό μια συνάντηση με την Επιτροπή στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ, κυρία Φαγά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κύριο Γιακολίνο για το εξαιρετικό του έργο αλλά και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι αυτό το έγγραφο ε, συμπεριλαμβάνει όλο το έργο που έχουμε υλοποιήσει με, όλες, με όλα αυτά τα θεματικά έγγραφα και άλλα κείμενα που προετοιμάσαμε κατά τη διάρκεια ε, της προετοιμασίας μας. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του ξεβλήματος νομικού χρήματος, ε, των ε, φορολογικών παραδείσων. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι δείχνουν το ύψος ε, των χρηματικών ποσών που χάνουν οι Ευρωπαίοι κάθε χρόνο. Και ιδίως εν μέσω κρίσης καθίσταται ακόμα πιο σαφές πόσο σημαντικό είναι να, πιο πόσο σημαντικό είναι να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα που σήμερα είναι ένα παγκόσμιο και όχι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο υπεύθυνη πολιτική, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, ε, στο δικαστικό σύστημα, στο έργο της αστυνομίας και άλλων αρχών. Και εφόσον εξετάζουμε τα στοιχεία που αφορούν τη διαφθορά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον χώρες όπου οι πολίτες μπορούν να πούν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αποτελεσματική. Επομένως, πλέον οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πια το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Προσωπικά θα ήθελα να προσθέσω ακόμα μερικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο και όταν μιλάμε για τον ρόλο του διαδικτύου. Στη σελίδα 8 λοιπόν, καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πρέπει να πούμε ότι το διαδίκτυο είναι μόνο ένα μέσο, ένα εργαλείο ε, το, το οποίο καταχράται το οργανωμένο έγκλημα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία κατά τη γνώμη μου του διαδίκτυο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Και βεβαίω πρέπει να ληφθούν και μέτρα κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όταν μιλάμε για την οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα της μαφίας, θεωρώ ότι ο εισηγητής πολύ συχνά αναφερόταν ε, ε, αναφερόταν στις οργανωμένες ε, ομάδες εγκληματιών και όχι τόσο στη μαφία. Πρέπει να υπάρχει μια σωστ... ένας σωστός διαχωρισμός μεταξύ των δύο. Απέναντίας σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, νομίζω ότι η έκθεση θα έπρεπε να ε, προβάλλει περισσότερο τη διαφθορά ως ε, μεμονωμένο φαινόμενο και όχι ως δίωδο ε, που αξιοποιούν ε, αυτές οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για να ε, επεκτείνουν την επιρροή τους. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερος ορισμός της διαφθοράς και να μεταβιβάσουμε ένα σαφές μήνυμα σε σχέση με τη διαφθορά. Γιατί η διαφθορά δεν συνδέεται μόνο με το δημόσιο τομέα, υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, για τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος, θα ήθελα να συμφωνήσω ε, με την προηγούμενη μιλήτρια σε ό,τι αφορά την αύξηση, την ανάπτυξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ε, που έχει ε, άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία των ε, κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εξίσου μεγάλη επίπτωση και αντίκτυπο έχουν και στα δημοκρατικά συστήματα και κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών. Εξάλλου, θα πρέπει ξεκάθαρα να ορίσουμε τις δραστηριότητας οργανωμένου εγκλήματος και τις ποινικέ πράξεις, αξιόπινες πράξεις. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όλες τις αξιόπινες ε, πράξεις. Μιλήσαμε και για τα, φαινόμενα ε, στον αθλητισμό Ε, μεταστημένα παιχνίδια που δεν συνδέονται οπωσδήποτε πάντα ε, με το ξέπλυμα χρήματος. Πολύ συχνά αυτές οι δραστηριότητες συνδέονται ε, με, με την εγκληματική πηγή των εσόδων αυτών και γι' αυτό θα πρέπει σε αυτό να συμμετάσχουν και οι παγκόσμιες, ε, οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες και να προβάλλουμε και το δικό τους ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Ούτως ώστε οι κυρώσεις ε, να βρίσκονται στο ύψος ε, των παράνομων αυτών εγκληματικών πράξεων. Παράλληλα, πρέπει ξεκάθαρα να ορίσουμε τη θέση μας σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, και, του, και το ρόλο τους ε, σε αυτόν τον τομέα. Αναφερθήκατε στη Europol, στη Eurojust. Όμως, η αποτελεσματικότητα αυτών των οργανισμών αντιστοιχεί ε, στο μέγεθος του φαινομένου. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δημόσιες προμήθειες που ε, χρησιμοποιεί ως κριτήριο μόνο την ελάχιστη ε, τιμή. Γιατί αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ε, επέκταση ε, φαινομένων διαφθοράς. Ήδη αναφέρατε και το έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Και βεβαίως ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά ε, τέτοια φαινόμενα διαφθοράς και εγκληματικών πράξεων. Μετά, σε ό,τι αφορά την επιτήρηση των αρχών που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία και της ερευνητικής δημοσιογραφίας, μάλιστα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να επεξεργαστούμε τον ρόλο των ε, μεγάλων ε, καναλιών όπως το CNN. Και τέλος, ένα πρόβλημα που συνδέεται με την ε, χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα, γιατί η απαγόρευση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων μπορεί να έχει επιπτώσεις αντίθετες σε αυτές που επιθυμούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν και γι' αυτό δεν θα ήθελα να στηρίξω αυτή την πρόταση. Ο πολιτικός ε, στόχος σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλήματος χρήματος. Αυτός ο πολιτικός στόχος λοιπόν θα πρέπει να υπερβαίνει την, ε, το διαχωρισμό μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας δυνάμεις μας και όλοι μαζί ε, να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στίχους και να υπερβούμε ε, τις πολιτικές μας διαφορές. διαφορές συγγνώμη. Αυτό θα ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό πολιτικό μήνυμα από πλευράς μας και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα που έχετε υποβάλει δεν έχω καμία αντίρρηση. ίσως θα μπορούσε αυτό το θέμα να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της ε, Ολομέλειας του Απριλίου, αυτό θα ήταν εξαιρετικά θετικό. Και μπορούμε έτσι να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νιούτον Ντάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλή για το ξεκίνημα. Πολλές τροπολογίες ε, θα υποβληθούν, πιστεύω εκατοντάδες. Εγώ προσωπικά θα υποβάλω 50. Έχω ορισμένε διαδικαστικές ερωτήσεις και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να έχουμε τις απαντήσεις. Ο κανονισμός λέει ότι θα έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης και μετά μια τελική έκθεση. Άρα αυτή είναι η ενδιάμεση το ενδιάμεσο σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από τη Γραμματεία ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τροπολογιών για την τελική έκδοση της έκθεσης ε, πριν από την υποβολή στην Ολομέλεια και πότε πρέπει να ψηφίσουμε. Ο κανονισμός ε, ε, μας κάνει υποχρεωτική την υποβολή, ζητάει δηλαδή μια ενδιάμεση και μια τελική έκθεση. Λοιπόν, ποια είναι η προθεσμία τροπολογιών για την προσωρινή έκθεση. Είναι η επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αν είναι την ερχόμενη Δευτέρα, ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Την 5η, 18 Απριλίου στο Στρασβούρο έχουμε μία συνεδρίαση για να εξετάσουμε τις τροπολογίες θα είναι στις 9 το πρωί, θα είναι το απόγευμα, μπορεί να, έχουμε, να μας ενημερώσει η γραμματεία. Όλα αυτά είναι διαδικαστικά. Και επίσης τι θα κάνουμε για την προθεσμία αποβολή τροπολογιών για την τελική έκθεση και την ψηφοφορία επί της τελικής έκθεση και της τροπολογίας για το Στρασβούργο και επίσης τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα για την προσωρινή έκθεση και το χρονοδιάγραμμα του Στρασβούργου. Θα ήθελα πληροφορίες παρακαλώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την τελική έκθεση, μου δείχνει η γραμματεία. Το σχέδιο έκθεσης θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 13 Μαΐου. Η θα γίνει η παρουσίαση στις 17 Ιουνίου και η, η προθεσμία για τροπολογίες θα είναι 27 Ιουνίου. Η πρώτη συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει 10-11 Ιουλίου. Ενδεχομένως θα γίνει μία έκτακτη συνεδρίαση για την δεύτερη συζήτηση των τροπολογιών. Ε, μπορεί να γίνει σε 9 Σεπτεμβρίου και η οθέτηση στις 17 Σεπτεμβρίου με το τρέχον χρονοδιάγραμμα για την ενδιάμεση έκθεση ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα για το Στρασβούργο ε, ε, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα. 9, το 9 η ώρα το πρωί. 9 με 10 και μισή. Και επίσης, λέει ο κύριος Νιούτον Ντάν, προθεσμοί υποβολή τροπολογιών για την ενδιάμεση έκθεση. 26, 26 Μαρτίου, 5 το απόγευμα λέει ο πρόεδρος, την τρίτη δηλαδή. 26 Μαρτίου. Ο πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γκόμες, πρέπει να πω ότι και εγώ πρέπει να φύγω για 20 λεπτά μετά τις 4 και 10. Θα ήθελα λοιπόν ή δυνατόν να έχουμε κλέξει τον ε, πρώτο αντιπρόεδρο μέχρι τότε. Είμαστε 11 μέλη αυτή τη στιγμή. Έναν, ένα μέλος χρειαζόμαστε για να κάνουμε την εκλογή. και να αναλάβει την ε, προεδρία. Μέλος ή αναπληρωματικό μέλος. Αλλιώς θα πρότεινα να κάνουμε μία δοκιμή με τη συνάδελφό μας, την μελλοντική πρώτη αντιπρόεδρο και την ρωτώ. Μπορείτε να αναλάβετε έστω δοκιμαστικά το ρόλο μου στις 4 και 10, αλλιώς θα πρέπει να διακόψω. Συμφωνούν οι συντονιστές. Εάν θέλετε, θα πρέπει να, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει απαρτία, έτσι δεν είναι, για να γίνει κάτι τέτοιο. Alors, euh, Κατανοώ ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί βάσει των κανόνων μας, ε, αλλά εφόσον ε, βρισκόμαστε και στο διαδίκτυο και είναι απολύτως δημόσια η συνεδρίασή μας, η γραμματεία μου λέει να μην ε, ακολουθήσουμε αυτή την οδό. But we have to follow the rules. Πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες. Ε, βεβαίως. Γιατί όμως δεν μπορούμε άτυπα να προτείνουμε στην ενδεχομένω μελλοντική πρώτη αντιπρόεδρο να κάτσει στην καρέκλα σας κύριε πρόεδρε, ακόμα και αν δεν έχει εκλεγεί επισήμω. Ναι, ακριβώς αυτό θα πρότεινα και εγώ λέει ο πρόεδρος για να μην χάσουμε 20 λεπτά για να αναγκαστώ να διακόψει γιατί είναι μια σημαντική συζήτηση για αυτή την ενδιάμεση έκθεση. Εάν συμφωνείτε λοιπόν θα μπορούσατε να αναλάβετε την Προεδρία και Ελπίζω... Α, έχουμε όμως την είδηση ότι ο κύριος Ταβάρες ε, έρχεται στην αίθουσα, θα είναι εδώ σύντομα και <clears throat> θα του ζητήσω να κάτσει στη θέση μου και ελπίζω η κυρία Γιώτοβα να συμφωνεί. This is what they call improvising, isn't it? Εδώ αυτό σχεδιάζουμε. Okay. We have a quorum. You're very welcome. You're very welcome. Um, then I can now go... Λοιπόν, ο πρόεδρος, επανέρχομαι τώρα στο σημείο που συζητάμε. Είναι το 4. Όλα λοιπόν βαίνουν καλώς. Στο, είναι το σημείο 4, εκλογή πρώτου αντιπροέδρου. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες έχουν προτείνει την κυρία Ιώτοβα. Έχουμε τώρα πάνω από 12 μέλη, έχουμε 13 και μπορούμε να ψηφίσουμε. Παρακαλώ, όσοι συμφωνούν με την εκλογή της κυρίας Ιώτοβα, σηκώσουν το χέρι. Σαφέστατα λοιπόν ε, εκλεγήκατε με ομοφωνία πρώτη αντιπρόεδρος της ομάδας, της ομάδας μας. you Είσαστε η πρώτη αντιπρόεδρος. Μπορείτε λοιπόν τώρα αμέσως να αναλάβετε την προεδρία. Έχετε ολοκληρώσει, κύριε Ευχαριστώ, κυρία Αντιπρόεδρε, για την εκλογή σας. Και ευχαριστώ και τον κύριο Γιακολίνο για την εμπεριστατωμένη του ε, έκθεση, το σχέδιο έκθεσης ε, που αποτελεί μια εξαιρετική βάση εργασίας για μας. Έχω μερικές ερωτήσεις. Καταρχάς, βλέπω ότι στην έκθεση δεν αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα. Έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή. Να μην αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα Why concrete cases... Και ε, αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει κάποιος ειδικό λόγος για τον οποίο δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα μπορούσαν αυτά να είναι χρήσιμα. Επειδή γενικά πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στην ουσία. Ε, θέλουμε όμως να δώσουμε ένα έντονο μήνυμα, ε, όχι να γράψουμε γενικότητες επί των οποίων όλοι θα συμφωνήσουμε και αναρωτιέμαι εάν ε, οι συγκεκριμένα παραδείγματα θα προσδώσουν μεγαλύτερη χρησιμότητα ε, στο σχέδιο έκθεσης. Συνεχία συνεχεία θέλω να τον ρωτήσω κάτι που νομίζω δεν αναφέρεται, τουλάχιστον εγώ δεν το πρόσεξα. Είναι το θέμα του παράνομου πλουτισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται στη Σύμβαση κατά της ε, διαφθοράς. Και αναρωτιέμαι αυτό το θέμα του παρανοπλουτισμού πλουτισμού αν μπορεί να συμπεριληφθεί, ε, διότι μας απασχολεί από πλευράς πολιτικής. Είναι ένα πολύ αντιφατικό και ε, φλέγον θέμα σε ορισμένες χώρες και σε ήθελα να το ρωτήσω εάν μπορεί να αναφέρει αυτές τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των κρατών μελών. Η τρίτη μου ερώτηση είναι η εξής. Αναφέρει το τραπεζικό σύστημα, το ξέπλυμα χρήματος και σημειώνω ότι ο κύριος Γιακολίνο μιλάει για τη σημασία της Ένωση των Τραπεζών ε, που προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Όμως δεν θα έπρεπε να αναφέρομαι σήμερα το ανταγωνιστικό σύστημα φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών. Είναι ένα σύστημα το οποίο ενθαρρύνει φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και, και εξέπλημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε και από αυτή την προοπτική. Και γι' αυτό ρωτάω τον συνάδελφο κύριο Γιακολίνο ποια είναι η απόψη του για την απόφαση που ελήφθη το περασμένο Σάββατο τώρα προχτές από το Eurogroup να επιβάλλει ένα κούρεμα σε όλες τις τραπεζικές καταθέσεις σε ένα κράτος μέλος μας στην Κύπρο με τη δικαιολογία ότι ότι η Κύπρος θεωρείται ε, ένα κέντρο ξεπλήματος παράνομου χρήματος για όλες τις εγκληματικές οργανώσεις, τις ρωσικές, τη μαφία, τις μαφιόζους κλπ. Και τον ρωτώ εάν είναι σωστό να φορολογήσει τους φορολογούμενους πολίτες της Κύπρου. Διότι είναι πανεύκολο για όλους τους μαφιόζους και εγκληματίες να πληρώσουν ένα 10% κάτι ψηλά δηλαδή και να διαιωνίσουν το όλη αυτή τη διαδικασία ξεπλήματος ε, χρημάτων. Ο κ. Διακολίνο είπε ότι αυτές δεν είναι και οι μόνες εγκληματικές οργανώσεις, έχουμε και άλλες. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κατά την άποψή του πώς κρίνει αυτή την εξέλιξη στην καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, και θα ήθελα να ακούσω την άποψή του μετά από τα τελευταία γεγονότα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κάποιος άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Κύριε Σκουλίνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και Ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ με τη σειρά Άκουσα όλες τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων της κυρίας ε, Βερονίκ Ματιέ, Τάνια Φαϊγιόν, του φίλου μου και τη συναδέλφου Γκόμες. Όλες οι παρεμβάσεις αποτελούν πλούτο, πλουτίζουν ε, τα στοιχεία που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαμε σε επαφή με όλους τους σκιώδεις στο Στρασβούργο. Συμφωνώ με τη Βερονίκ Ματιέ όταν ε, μιλεί για συμφωνίες με τρίτες χώρες για την ανακύκλωση του βρώμικου χρήματος και τους φορολογικούς παραδείσους και βεβαίως ο θάνατος και η φτώχεια σχετίζονται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα. Θα δούμε κατά πόσο στο Στρασβούργο θα ασχοληθούμε ε, με το θέμα μέσω συντονιστών. Ίσως εκείνη τη στιγμή θα ορίσουμε καλύτερα το ζήτημα. Η συνάδελφος Φαγιούν αναφέρθηκε στην προαπέτηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης και συμφωνώ και εγώ ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να υπάρχει για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είμαστε ε, πεπισμένοι ότι και το έγκλημα στον ε, κυβερνοχώρο αυξάνεται. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τη ε, διαφθορά και πώς θα μπορέσουμε να διασαφίσουμε καλύτερα έναν ορισμό ο οποίος δεν είναι ε, σαφής. Για, ως προς τα match fixes είπαμε ότι θα αντιμετωπιστούν και βεβαίως ε, και η χρήση χρημάτων παράνομης προέλευσης είναι ένα φαινόμενο που όλο ένα και διαστέλλεται και αφορά και τον αθλητισμό γενικότερα. Τώρα, πώς μπορούμε να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο καλύτερο, σαφέστερο. Έτσι ώστε η προσφορά στις δημόσιες προμήθειες, η προσφορά να εγκρίνεται με βάση το δημόσιο συμφέρον. Αυτός να είναι ο γνώμονας. Θεωρούμε ότι ο, ως προς την ε, ε ακτοπλοεία και την ακτοφυλακή θα πρέπει να αρκεστούμε στο Eurojust και στη Europol. Η κυρία Φουαγιόν ίσως θα μπορούσε να μας πει ε, πού ακριβώς αναφέρεται. Ο συνάδελφος Νιούτον Ντάν μίλησε για τις διαδικασίες και για τις απαιτήσει που διαγράφονται εκ των προτέρων, όπως είπε και η Βερονίκ Ματιέ. Εγώ σας έδωσα ορισμένες χρονικές ενδείξεις, γνωρίζοντας ότι στις 18 Απριλίου μπορούμε να συναντηθούμε στο Στρασβούργο. Ας βρούμε μια λύση που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα. Όπως ξέρετε, Στην περίπτωση του Στρασβούργου ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μία μεγαλύτερη και αθρώα προσέλευση των συναδέλφων. Εν πάση περιπτώσει μπορώ να δεχτώ και διαφορετικές εναλλακτικές. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Φαγιόν όταν μίλησε για χρηματοδότηση των κομμάτων. Θα πρέπει να μην γίνεται διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Η συνάδελφος Γκόμες υπέβαλε μια σειρά ερωτήσεων. Ας αρχίσουμε από την πρώτη γιατί δεν αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα βλέπετε στις μεμονωμένες εκθέσεις ότι βασιστήκαμε στα θετικά εθνικά νομοθετικά στοιχεία. Άρα Ξέρουμε ότι στην περίπτωση της Δανίας υπήρξε, έγινε ειδική πρόοδος ως προς το ελεγκτικό συνέδριο. Αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα εθνικά πλαίσια για να μιλήσουμε για μία βάση ευρωπαϊκής προσέγγισης ως προς τη διαφθόρα. Είμαστε υπέρ κοινών νομοθετικών πλαισίων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά με συγκεκριμένες αυστηρές ε, κυρώσεις. Μας ενδιαφέρει η θέση των πολιτικών. Ως προς το θέμα του ξεπλήματος, μιλήσαμε για την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των τραπεζών που είναι πιο υπεύθυνες και αυτό μαζί και με τους συμβολεογράφους που θα μας βοηθούσαν να εξηχνιάσουμε ή να ανοιχνεύσουμε ε, επίμαχες ή ύποπτες πράξεις. Δεν υπάρχει βεβαίως ε, πλήρης εξισορρόπηση στα κράτη-μέλη ως προς την απάτη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Το έγγραφο αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές ε, για να είμαστε πιο υπεύθυνοι, να είναι πιο υπεύθυνα τα κράτη-μέλη και να μπορέσουν πιο αποδοτικά να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Βεβαίως ε, υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Κύπρος, που αντικειμενικά, όπου αντικειμενικά υπάρχει μία ήπια αντιμετώπιση ε, ως προς το ξέπλυμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο αλλού φορολογική παράδοση. Παραδεισί. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί για να επανευθυγραμμίσουμε τη γραμμή των κρατών μελών. Σύμφωνα με την κυρία ε, Γκόμες επί του θέματος. Και ο Επίτροπος Σεμέτα βρέθηκε εδώ μεταξύ μας και μας μίλησε για μία ε, φορολογική και δημοσιονομική πολιτική όπου θα ενταχθεί και η τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματος. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για φορολόγηση με 10% των ε, καταθέσεων και το θέμα αυτό είναι επίμαχο, δεν ξέρουμε ε, κατά πόσο είναι απόλυτα νόμιμο. Είναι διφορούμενο. Τέλος, ε, θα ήθελα να πω ως προς τα διαδικαστικά ότι εμείς υποβάλαμε μία πρόταση από κοινού με τη γραμματεία που προβλέπει η προθεσμία υποβολή στις 26 και όχι 25 για να έχετε άλλη μια μέρα στη διάθεσή σας. Είμαι πεπισμένος ότι οι ομάδες ε, συνεισέφεραν και με επιμέρους συνεισφορές και θα μπορούσαμε να προβάλλουμε ένα κοινό project όπως τα κρίνει και ο εισηγητής. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Απριλίου γιατί το πρόγραμμά μας θα οριστεί από κοινού με τους συντονιστές. Θεωρούμε ότι το Μάιο ή τον Ιούνιο θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε την ενδιάμεση έκθεση η οποία μας απασχολεί σήμερα. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Άρα σας ξαναδίνω το λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Η γραμματεία προβλέπει άλλο. Έχει προβλέψει κι άλλο ένα θέμα για τη συνάντησή μας. Πρόκειται για την έκθεση της επίσκεψης της αντιπροσωπείας μας στη Χάγη αλλά δεν βλέπω εκπροσώπους. Γι' αυτό διακόπτουμε και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών στην έκθεση για, το, για Κολίνο είναι στις 26 Μαρτίου στις 5 ε, το απόγευμα. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις, διακόπτουμε μέχρι τις 17.30. Οι συντονιστές θα συναντηθούν στις 5.30. Σας ευχαριστώ.